αφού κάναμε την αναδιάρθρωση εδώ στις Καράκλες, για να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Πάρτε θέσεις. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα σημαντικά και σημαντικά σημεία στη μέση διάταξη. Καταρχά, έχουμε τη μελέτη σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και το πρόγραμμα καινοτομίας Ο Πάολ Ρούμπιχ είναι ο εισηγητής, ο οποίος ασχολείται πολλά χρόνια με, την, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι γνωστός στους κύκλους αυτούς. Και επίσης εδώ να καλωσορίσουμε την κυρία Τόντλινγκ Σιονχόφα και την κυρία Μπάουερ που θα μας κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Παρακαλώ, Πάολα, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, να ευχαριστήσω που ε, κατέστη δυνατόν να γίνει αυτή η μελέτη, γιατί η ανεργία στην Ευρώπη ε, είναι ο βασικός στόχος για την ε, υπερχρέωση των κρατών και αυτό φαίνεται όχι μόνο από το τι θα γίνει στο μέλλον με τις επιχειρήσεις, αλλά το, με το, σχετικά με το πώς μπορεί κανείς ανεξάρτητα να εργαστεί, πώς ε, μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η ανεξαρτησία των εργαζομένων και τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος ε, είναι αυτοαπασχολούμενος και ε, προσλαμβάνεται κάπου. Υπάρχει το πρόγραμμα SIP, πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία, για να προωθηθούν όλες αυτές οι επιτυχίες. Πρέπει να δούμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα, τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος. Για μας το πρόγραμμα αυτό είναι μια πολύ σημαντική βάση για να μπορέσουμε να κρίνουμε από τα προγράμματα ε, για τις ε, μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει τώρα και για τα οποία το Κοινοβούλιο έχει δώσει 5 δισεκατομμύρια. Στο ΣΥΠ δώσαμε 3,8 και το ε, Συμβούλιο προτείνει 2,03 δις. Σημαντική μείωση δηλαδή. Γι' αυτό θεωρώ ότι για το Κοινοβούλιο είναι να δούμε πώς μπορούμε το ε, πρόγραμμα αυτό να το δομήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο, πώς μπορούν οι επιχειρήσεις μέσω πρόθεσμα, ε, ε, βράχη πρόθεσμα συγγνώμη, να λαμβάνουν αποφάσεις και πώς μπορούν να εισραίουν τα κονδύλια στις επιχειρήσεις αυτές. Επίσης, η αξιολόγηση του προγράμματος ΣΥΠ είναι πολύ σημαντική για το Κοινοβούλιο και ευχαριστώ που μέσα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε με αποτελεσματικό και καλό τρόπο να αναλύσουμε την κατάσταση. Ε, θα περιμένω να ακούσουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Τόντλινγκ Σιενχόφα. Σύντομα και γερμανικά θα μιλήσω. Χαίρομαι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τόσο συναρπαστικό θέμα. Έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά ε, αξιολογήσεων, αλλά έχουμε κάνει πέντε μετααξιολογήσεις, δηλαδή αξιολογήσεις αξιολογήσεων. Και ποιο είναι τώρα το αποτέλεσμα το οποίο έχει ε, προκύψει. Οι αξιολογήσει έχουν καταδείξει πόσο κατακαιρματισμένο είναι το πρόβλημα αυτό και πόσο πολυσχηδές στις επιδιώξει του. Όλα αυτά τα κάναμε στα αγγλικά βέβαια. Και ο συνάδελφός μου που έχει συμμετάσχει στην έρευνα θα κάνει αυτή την μεταξιολόγηση στα γερμανικά. Γιατί είναι δύσκολο να γίνεται αυτή η ε, εργασία στα γερμανικά. Η κυρία Μπάουερ λοιπόν. Ωραία. Ναι, στα γερμανικά ευχαριστώ και τώρα θα τα πω αγγλικά. Είναι χαρά μου που μπορώ να παρουσιάσω σήμερα στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Θα ήθελα να τη διατρέξω. Θα κάνω μια επισκόπηση αρχικά της παρουσίασής μου και εν συντομία θα παρουσιάσω τους σκοπούς, πώς διοργανωθήκαμε, πώς διοργανώθηκε η όλη διαδικασία μαζί με τους διάφορους εμπειρογνώμονες που είχαμε και να σας θυμίσω εάν το αμελήσατε, τι είναι το SIP και το AIP, Δηλαδή, το πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Θα σας πω τι κάναμε στην μελέτη, ποιες ήταν τα βασικά, τα βασικά ευρήματα και ποιες οι συστάσεις μας. Έχει δύο τμήματα η μελέτη. Το ένα αφορά το πρόγραμμα SIP, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, και το άλλο τα λειτουργικά προγράμματα τα ΙΑΕΠ, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Μετά θα μπούμε στην ουσία της ε, μελέτης που αφορά τι συστάσεις. Υπάρχουν 22 συστάσεις στη μελέτη και θα προσπαθήσω να τις διατρέξω σύντομα για να καταλάβετε τι έγινε. Ποιος ήταν ο σκοπός της μελέτης. Όπως προείπε η συνάδελφος, δεν είχαμε μια πραγματική επιτυχία τόπια αξιολόγηση ήταν μια μεταξιολόγηση θεωρητική, ειδικά για το ΣΥΠ. Πήραμε τις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν γίνει ως τώρα, αυτό ήταν το πρώτο τμήμα και μετά παίρναμε ένα λειτουργικό πρόγραμμα, το EIP, το εμπαθύναμε και βλέπαμε ποια ήταν τα ωφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσπαθώντας να αντλήσουμε συμπεράσματα. Για να ξέρετε πώ διοργανωθήκαμε από την πλευρά του χρονοδιαγράμματος, ξεκινήσαμε πέρσι τον Οκτώβριο που συναντηθήκαμε στο Κοινοβούλιο και ξεκινήσαμε τότε την έκθεση αποτίμηση. Assessment report. Για να έχουμε πραγματική αξιολόγηση των διαφόρων εκθέσεων. Εάν ξέρατε το πρόγραμμα, θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλέ εκθέσει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκθέσεις αξιολόγησης και αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης ετοιμάζονταν από τρεις ε, εμπειρογνώμονες της ε, εκτίμησης ομοτήμων ήδη από τον Οκτώβριο. Τρεις λοιπόν οι ειδικοί, ανεξάρτητοι και τρεις, όπου τελικά αυτή η διαδικασία οδήγησε σε μια συνάντηση τον Νοέμβριο για να φτάσουμε σε συμπεράσματα μαζί με την βασική ομάδα και τους τρεις εμπειρογνώμονες που είχαμε επιλέξει και βάσει των συμπερασμάτων αυτή της συνάντησης και κάποια ε, μελέτη της βιβλιογραφίας καταλήξαμε την ολοκλήρωση της έκθεσης το 2012 και την περάτωσή της το Μάρτι φέτος. Αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα. Ήταν εντατικό το πρόγραμμα. Να σας θυμίσω για το SIP, πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Είναι πολλά τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. Είναι μια δομή που θα ολοκληρωθεί το 2013. Διοργανώνεται, διαρθρώνεται καλύτερα σε, τρεις, σε τρία λειτουργικά προγράμματα. Το ένα είναι το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία δηλαδή συνεργασία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτά, σε αυτές είναι ανοιχτό, ενώ τα υπόλοιπα σε όλων των ειδών της δομές και οργανώσεις. Ένα είναι αυτό για τις ε, τεχνολογίες ε, πληροφορίας και επικοινωνιών και το άλλο για την ευφυή ενέργεια στην Ευρώπη. Μας απασχόλησε κυρίως το ΙΑΕΠ με 2.170 εκατομμύρια και 720 εκατομμύρια για τα άλλα δύο προγράμματα. Για το μέλλον τώρα. Ξέρετε ότι υπάρχει μεταβατική περίοδος. Το ΣΥΠ και, το πρόγραμμα πλαίσιο 7 θα ολοκληρωθούν και θα λήξουν το 2013. Πολλά πρέπει να γίνουν ώστε να ετοιμάσουμε την πορεία για τα επόμενα προγράμματα, το πρόγραμμα Horizon και το COSME. Φαίνεται ότι πολλές συζητήσεις γίνονται ήδη για τον προπολογισμό και το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων. Ποια ήταν τα συμπεράσματα, τα βασικά ευρήματα από τη μελέτη των εκθέσεων. Πρώτα απ' όλα, συμπεράσματα για την αξιολόγηση του ΣΥΠ. Οι εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν εκπονηθεί ως τώρα για το πρόγραμμα ΣΥΠ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενδιάμεσες εκθέσεις και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης για το πρόγραμμα ΣΥΠ και για τα τρία λειτουργικά προγράμματα από διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές οργανώσεις. Αυτό που βρήκαμε ήταν και προφανές είναι ότι το πρόγραμμα διαιρείται σε τρεις βασικές δραστηριότητες μη συγκρίσιμες. Με διαφορετικούς στόχους, οι δύο είναι ε, με διαφορετικό περιεχόμενο και με άνοιγμα σε όλους τους δικαιούχους. Είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε το συνολικό αντίκτυπο του προγράμματος ΣΥΠ, γιατί ακριβώς υπάρχει τέτοια ετερογένεια. Το επόμενο στοιχείο Έτσι όπως το είδαν μάλιστα οι εμπειρογνώμονες, είναι ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος ΣΥΠ και των λειτουργικών του προγραμμάτων ήταν γενικώ καλής ποιότητας, όμως και πολύ ετερογενή ως προς την μεθοδολογία, ενώ η περίοδος που πέρασε μεταξύ της ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης ήταν 20 μήνες κατά μεσόρο η τελική έκθεση δεν είναι τελική στην πραγματικότητα, απλώς δίνει πληροφορίες για το 60% των ενδιάμεσων προγραμμάτων ή το πρόγραμμα SIP. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο. Εάν δούμε τώρα τις συστάσεις, βλέπετε και τα συμπεράσματά μας. Επιπλέον τον οσον είπα, η ειδική ομότιμη αξιολόγησης είδα ότι χρησιμοποιείται διαφορετική ορολογία ω προ τους δείκτε. Κάποιες φορές υπάρχουν σοβαρέ αποκλήσει. Η προσέγγιση των δικτών είναι γενικώ πολύ περιπλοκή και υπάρχει μεγάλο περιθώριο για απλούστευση. Αυτή η συζήτηση μάλιστα γίνεται ήδη και είναι σε εξέλιξη και για άλλα προγράμματα και άλλα πολιτικά εργαλεία. Αυτά ήταν τα βασικά ευρήματα για το ΣΥΠ και την αξιόλογη, από την αξιολόγησή του. Τώρα, συγκεκριμένα στοιχεία για τα χρηματοδοτικά μέσα του EIP. Κάτι που ενδιέφερε ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο, γι' αυτό θα σταθώ εδώ. Βασικά ευρήματα λοιπόν. Βασική κατηγορία δικαιούχων, μικρομεσαίες επιχειρήσει με λιγότερου από 10 εργαζομένου και 100.000 ετήσιο τζίρο. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία απέδιδαν 53% του προπολογισμού για διάφορα μέσα, τα οποία κάλυπταν τις ε, εκτελούνταν, μάλλον ε, χρησιμοποιούνταν τα πανόντα πλήρως. Ειδικαίως τώρα για τα GIF, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με υψηλή ανάπτυξη και ιδιαίτερα καινοτόμες. Υπήρχε χρηματοδότηση και με αξιόγραφα και για άλλες ειδικέ δραστηριότητες παρατηρήσαμε ότι οι δικαιούχοι είναι κυρίως άρενες. Εκτός από τις μικροπιστώσεις που σε μεγάλο βαθμό απευθύνονται και σε γυναίκες δικαιούχους. Γενικώ, το πρόγραμμα EIP καλύπτει ένα φάσμα διαφορετικών υπηρεσιών. Αν ρίξετε μια ματιά στην επόμενη σελίδα θα δείτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πολλά ε, μέσα στήριξης πολιτικής, θεματικές δραστηριότητες, εσωτερικές δραστηριότητες, πολλά στοιχεία και αυτό κάνει την αξιολόγηση πολύ δυσχερή. Γιατί κάθε δραστηριότητα διαφέρει πολύ από, την, ε, από μια άλλη. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσουν στι συστάσει. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια ευθυγράμμιση, κάποιο εξοδολογισμό στο μέλλον. Επί τη αρχή ενδιαφέρονταν όλοι βάσει τη μελέτη μα για την δημοσίευση πληροφοριών το πρόγραμμα για την ε, πληροφορία και τις τεχνολογίες της ε, δίνει πολλά στοιχεία για την καινοτομία, τις εξελίξεις. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, ενώ το δίκτυο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ήταν ε, ιδιαίτερα επιτυχές με θετικές αποκρίσεις από τους χρήστες. Αυτά ήταν τα βασικά ευρήματα. Ας έρθουμε τώρα στις συστάσεις. Εάν διατρέξετε τη μελέτη μας, θα δείτε ότι έχουμε 22 συστάσεις Προσπαθήσαμε να τις ομαδοποιήσουμε κάπως για να μπορείτε κι εσείς να καταλάβετε τι γίνεται. Ως προς τις εκθέσεις, νομίζουμε ότι οι ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης είναι πολύ κοντά χρονικά. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να γίνει μια προσπάθεια για να υπάρξει απόσταση μεταξύ των δύο σταδίων και να υπάρχει καλύτερη συνολική αξιολόγηση του αντικτύπου των προγραμμάτων. Υπάρχει πλούτος πληροφοριών στις διάφορες εκθέσεις, εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ε, προγραμμάτων της ε, εκτέλεσης, των επιδόσεων, της αξιολόγησης. Κάποιες φορές είναι αρκετά δύσκολο ιδίω ό,τι αφορά τον προπολογισμό και την επισκόπηση του, να θέσει κάποιο τα όρια. Υπάρχουν αποκλήσει μεταξύ των εκθέσεων ασυνέπειε, α το πούμε έτσι, κάτι που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, να βελτιωθεί στο μέλλον. Επιπλέον, εάν αποφασίσει κανεί να κάνει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγηση και τελική έκθεση αξιολόγηση, πολύ κοντά από χρονική άποψη, τουλάχιστον να σε ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία ή ας ε, χρησιμοποιεί την ίδια ομάδα. Ας βρει κάτι συγκρίσιμο. Διότι αυτό δεν συνέβαινε στην πράξη με τη μεθοδολογία ούτε με την ομάδα των δεδομένων που συγκρίνονταν. Αυτό ό,τι αφορά τι εκθέσει. Οι δείκτε τώρα. Οι δείκτε συζητώνται διαρκώ. Είναι μια ιστορία χωρί τέλο. Παρόμοιες συζητήσεις για τους δείκτες γίνονται και σε άλλα γενικά, σε άλλες γενικές διευθύνσεις, αλλά νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός με, τα άλλα, με τις άλλες γενικές διευθύνσεις. Ως προς το τελικό σύνολο των δικτών, η προσέγγιση θα μπορούσε να απλουστευτεί, θα έπρεπε να απλουστευτεί με συγκεκριμένη συγκεκριμένε οδηγίε για τον ορισμό των δικτών και ήδη από την αρχή λειτουργία του προγράμματος θα πρέπει να υπάρχει ένα βασικό σύνολο εμ, δικτών οδηγών ώστε να μπορούν όλοι να έχουν κατευθείαν μια συνολική εικόνα και να υπάρχει μια ρεαλιστική αποτίμηση του προγράμματος ε, ανατακτά χρονικά σημεία. Οι ειδικοί έδωσαν την εξή ιδέα. Να έχουμε τρία διαφορετικά επίπεδα για τους δείκτες. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μακροπρόθεσμους δείκτες, μακροοικονομικούς δηλαδή, που να απηχούν τους στόχους του προγράμματος. Μολονότι οι ειδικοί επεσήμαναν ότι πρέπει να το σκεφτούμε εάν τέτοιοι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιούνται και να, γίνουν, να κάνουν ε, ρεαλιστικές μετρήσεις. Εάν είναι εφικτό να τους χρησιμοποιούμε και να μας δίνουν τα αποτελέσματα που θέλουμε. Σε επίπεδο προγράμματος τώρα πρέπει να μετράμε το αποτέλεσμα και το, και το προϊόν, δηλαδή input και output. Και το αποτέλεσμα. Εδώ θα ήταν χρήσιμο να έχουμε δείκτες που σε επίπεδο εταιρεία ή τέλο πάντων δικαιούχου δείχνουν την εξέλιξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, εάν υπήρξε αντίκτυπος στη συγκεκριμένη ε, μικρομεσαία επιχείρηση από τη λειτουργία του προγράμματος. Αυτά για τους δείκτες. Τώρα για το πρόγραμμα, για τα προγράμματα σε αυτό το επίπεδο. Όπως είπα, είδαμε ότι οι μεγάλες διαφορές και ο περίπλοκος χαρακτήρας των προγραμμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί Πρέπει να υπάρξει ο εξορθολογισμό. Επίση, πρέπει να υπάρξει διασύνδεση με άλλε δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια, τη συνοχή και την πολιτική τη και τα εργαλεία που αυτή χρησιμοποιεί. Περιφερειακοί και τοπικοί παράγοντε μπορούν να αναλάβουν αυτή την υλοποίηση σε συγκεκριμένου τομεί, όπω τι δραστηριότητε εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Τεχνολογία και την Καινοτομία, καθώ και το δίκτυο για τι επιχειρήσει τη Ευρώπη. Και εκεί πρέπει να υπάρξει συντονισμός. Θετικά είδαμε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως τα help desk, τα γραφεία βοήθειας και τις δραστηριότητες διαδικτύωσης που βάσει της απόψης των ειδικών θα πρέπει να συνεχιστούν. Η... Η εβδομάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κάτι που θα μπορούσε να εξακολουθήσει και άλλες πρωτοβουλίες όπως το επιχειρήν για τις γυναίκες παρόλο που παραμένουν και κάποια προβλήματα. Επίσης θα μπορούσε να γίνεται διαφορετική αποτίμηση των τομεακών δραστηριοτήτων. Υπήρχαν πολλές ανατομέα όπως για τον τουρισμό, τον κατασκευαστικό. Θα άξιζε τον κόπο να γίνει αξιολόγηση για τον αντίκτυπο των δράσεων αυτών. Θέματα που έχουν να κάνουν με τις ίδιες τεχνικομεσαίες επιχειρήσεις τώρα, πιο συγκεκριμένα. Εάν δούμε μια μικρομεσαία επιχείρηση, πρέπει να πούμε ότι είναι φοβερές οι διαφορές ως προς το μέγεθος, το μηχανικό κλάδο, τι δυνατότητε έρευνα τη ίδια της επιχείρηση, τον κύκλο ζωής της και τη φάση στην οποία βρίσκεται. Η ιδέα των ειδικών, λοιπόν, η ιδέα που μας έδωσαν ήταν να κάνουμε καλύτερη ομοδοποίηση βάσει κάποιων ε, ειδικών χαρακτηριστικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ή τις ίδιες τις δραστηριότητες. Κάτι άλλο ήταν ότι θα ήταν συνετό να γίνει μια μελέτη ιδίω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή να επικοινωνήσουν, αλλά εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Να έρθουν σε επαφή με χρηματοδοτικά μέσα. Το θέμα είναι γιατί δεν προχωρούν. Θέλουμε και αυτό να το κρίνουμε. Επίσης, η χρονική απόσταση μεταξύ έγκρισης και την πραγματική λήψη της πίστοσης των κονδυλίων, αυτό δεν καταγράφεται στις εκθέσεις αξιολόγησης και μπορεί αυτό να δυσκολεύει συνολικά την ε, άντληση ωφελών από τα προγράμματα. Τέλος, οι εμπειρογνώμονες επέμειναν ότι πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα εργαλεία για την χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να ασχολούνται περισσότερο με την κάλυψη των κινδύνων. Και προφανώς θα γίνει συζήτηση και το συνδυασμό κάποιων προγραμμάτων με το Horizon 2020 το κόσμο, αυτή και η διαχείριση θα πρέπει να ρυθμίζεται ξεχωριστά από άλλο ρυθμιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή τέλος πάντων να συγκεντρωθεί σε ένα κοινό πρόγραμμα ώστε να αποδεχθούν προβλήματα. Αυτές ήταν οι διαφορετικές συστάσεις βάσει τις μελέτες μας. Τώρα είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπάουερ για την παρουσίαση της τόσο ενδιαφέρουσας έρευνά σα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στην Επιτροπή μας μάλλον, την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, στα μέλη της Επιτροπής μας. Ποιος έχει ένα ερώτημα ή κάποιο σχόλιο για αυτά τα οποία ακούσατε. Υπάρχει μια σωρία προτάσεων εδώ από τη δική σας πλευρά βλέπετε θετικά ή αρνητικά τις προτάσεις αυτές. Παρακαλώ. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο. Πράγματι χαιρετίζουμε ιδιαίτερα αυτή την έκθεση, η οποία περιέχει πολλές χρήσιμες <clears throat> συστάσεις για το πρόγραμμα. Χαιρόμαστε βλέποντες ότι πολλές από τις προτάσεις ευθυγραμμίζονται με τα πορίσματα της Κομισιόν από τις διάφορες ε, αξιολογήσεις για τα προγράμματα του CHIP. Του CHIP, Η θέση της Κομισιόν έχει παρουσιαστεί εν συνόψη σε έγγραφα προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών, την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 15 Ιανουαρίου 2013. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση μεταξύ της ανάγνωσης και των αξιολογήσεων της ε, Κομισιόν και των μετα, μεταξιολογήσεων αυτής της μελέτης. Και τα δύο έγγραφα αναγνωρίζουν πράγματι ότι ο, το πρόγραμμα SIP, ο πυλώνας αυτός για την ανταγωνιστικότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικός και αν δούμε την τελική αξιολόγηση, είναι φανερό ότι τα απορίσματα της τελικής αξιολόγησης είναι το SIP από αφεαυτού και τα επιμέρους προγράμματα λειτουργούν πολύ θετικά και καλύπτουν τις προσδοκίες. Και το ΣΥΠ είναι ένας να προωθήσουμε την καινοτομία. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν συμφωνούμε με τις συστάσεις που προέρχονται από αυτή την έρευνα. Αν μπορώ να πω κάτι για το, χρονισμό αυτής της ε, αξιολόγησης, προφανώς αυτό καθορίζεται από τη νομική βάση, αλλά έχετε μια επιλογή. Ή μπορείτε να έχετε μια πραγματική τελική αξιολόγηση όταν όλα ή σχεδόν όλα από τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα τρίχατε πολύ αργά στην διαδικασία. Αν είχαμε αυτή την αξιολόγηση το 2013 τότε ε, τελειώνει η περίοδος για τις ε, δεσμεύσεις πιστώσεων αλλά το EIF έχει ακόμα δύο χρόνια να συνάψει συμφωνίες και να δώσει εγγυήσει προς τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορεί να καλύπτουν πολυετή χρονικά διαστήματα. Επομένως, ε, αυτό θα ήταν λιγάκι καθυστερημένο. Εδώ η επιλογή ήταν να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούμε πριν εκπνεύσει το πρόγραμμα ώστε να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε το επόμενο πρόγραμμα, αυτό που σπάσει να κάνει και η Κομισιόν και πολλές από τις συστάσεις αυτές εφαρμόζονται ήδη στον τελευταίο χρόνο εφαρμογής του ΣΥΠ αλλά πολλά άλλα θα βρεθούν και στην πρόταση της Κομισιόν για τα νέα προγράμματα. Και αν δούμε την πολυπλοκότητα των προγραμμάτων αυτών που αποτελούν ένα σύμπλεγμα αλλά έχουν διαφορετικούς στόχους, μπορούμε να πούμε ότι στην πρόταση της επομένης περίοδου πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών αλλάζει κάπως η προσέγγιση. Θέλουμε να σωματώσουμε την καιροτομία στο ορίζοντα 2020 και θέτουμε περισσότερο στον πυρήνα την ανταγωνιστικότητα για τα πρόγραμματα αυτά. Για τους δείκτες, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό σύμπλεγμα θεμάτων. Είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία ε, τα είχαμε στη διάθεσή μας ήδη από την ενδιάμεση αξιολόγηση. Κάναμε μία και χωρισμένη <clears throat> αξιολόγηση για τους δείκτες και τώρα προχωρούμε στην εφαρμογή του προγράμματος COSME βασιζόμαστε σε αυτό το σύνολο δικτών για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε ένα πλαίσιο αξιολόγησης για τον κόσμο που θα μας βοηθήσει στο επίπεδο εφαρμογής. Θα περάσουμε λοιπόν από το επίπεδο δράσης στο επίπεδο εφαρμογής. Και σε ό,τι αφορά και τη νομική βάση, τις νομικές βάσεις, έχουμε ένα συνεκτικό σύνολο που θα έχουν ε, εφαρμογή σε τεχνικό επίπεδο και νομίζω ότι η Κομισιόν είναι πλήρης εμπιστοσύνη σε ότι έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο για την εφαρμογή. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες των συστάσεων αυτών, διότι θα μακρηγορήσω υπερβολικά. Απλώς θα ήθελα να αναφερθώ στην τελευταία παράγραφο της έκθεσης της Κομισιόν που προανέφερα, που προσκαλεί το Συμβούλιο, αλλά και το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσουμε πλήρως αυτή τη σύσταση όταν τροποποιούν την πρόταση της Κομισιόν ενώπιση της τελικής έγκρισης των προγραμμάτων και είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση γιατί βρισκόμαστε στις τελευταίες φάσεις της έγκρισης. Ευχαριστώ πολύ λέω πρώτος για τη θέση της Κομισιόν. Υπάρχει από την πλευρά της Επιτροπής μας κάποιος ο οποίος θέλει να αυτό, ο κ. Ρούμπικ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το γεγονός ότι αυτή η αξιολόγηση και μεταεξιολόγηση έλαβε χώρα. Πιστεύω ότι στο Κοινοβούλιο τώρα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του προγράμματος αυτού εν ώψη τη χρονική ε, περίοδου 2014-2020. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν του συντάκτε αυτή τη έκθεση. Ευχαριστούμε. Κυρία Τέρντλιχ, θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Θα ήθελα να να κάνω μια παρατήρηση στην πολιτική συνοχή. Υπάρχουν σημαντικά ποσά τα οποία χρησιμοποιούνται για τους στόχους αυτούς και από την πλευρά της Κομισιόν προβλέπεται ένα ποσό 8,9 ε, δισεκατομμυρίων, από τα οποία 1,2 αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε στην επόμενη χρονική περίοδο να βρούμε τις κατάλληλες συνέργειες και την σωστή οριοθέτηση των ενεργειών αυτών, ώστε να έχουμε μια παράλληλη ε, λειτουργία αυτών των εργαλείων. Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον τριγωνικό διάλογο, τον τριμερή διάλογο, τα θέματα συνοχής. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε το πώς είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε τη σωστή χρηματοδότηση για αυτά τα προγράμματα, αλλά ξέρω και για την Κομισιόν αυτό είναι σημαντικό θέμα και με, τον, με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων, ο κύριος Ρούμπικ και εγώ, θα είμαστε σε επαφή για να εξασφαλίσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ για τις τόσο ενδιαφέρουσες σκέψεις. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο διερευνήσατε και στο παρελθόν ο συνάδελφός μου ο κύριος Χαζημαρκάκης, το έχει αντιμετωπίσει με, κάποια με κάποιο σκεπτικισμό σε σχέση με την λυσιτέλεια του προγράμματος αυτού αν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία υπόσχεται, αλλά νομίζω ότι βάσει τη έκθεσή σα βλέπουμε ότι υπάρχουν αξιοσημείωτα θετικά αποτελέσματα και ω εκ τούτου είμαι πεπισμένο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας θα πρέπει να υποστηριχθούν με τον τρόπο αυτό και έχουμε παραγωγικά εταιρείε όπως η ASAP η εταιρεία πληροφορικής της Γερμανίας για τη νέα οικονομία. Έχουμε πολλές ε, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στον τομέα αυτό. Ξέρουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του σήμερα μπορεί να είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις του αύριο και ως εκ τούτου έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε. Θέλει να λάβει κανείς το λόγο, βλέπω όχι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνάς σας και όποιος έχει περαιτέρω ερωτήσει μπορεί να έρθει πάντα σε επαφή μαζί σας. Ευχαριστώ. Oh, Προχωρούμε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε λίγο μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το επόμενο σημείο λοιπόν είναι η σχετική μελέτη για τις δυνατότητες αναδιοργάνωσης του έργου ΙΤΕΡ με στόχο να βελτιωθεί η σχέση κόστους αποτελεσματικότητας. Πρέπει να προετοιμάσουμε λιγάκι τώρα εδώ την παρουσίαση. So, we... Okay. Um... Λοιπόν, να δώσουμε τον ε, λόγο στον ε, εισηγητή αν τον επιθυμεί. Κύριε Γκάιερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι. Ως ελεγκτές του προπολογισμού έχουμε ασχοληθεί ενεργά και στο παρελθόν με το θέμα του ΙΤΕΡ ανεξάρτητα βεβαίως από τα τεχνολογικά προγράμματα θεωρήσαμε ότι, το, ότι υπήρξε μεγάλο η άνοδος του κόστου, του κόστους για το ίτερ, όπου το ίτερ ε, από ένα απλό έτσι, πρόγραμμα ε, επιχάρτου έγινε ένα πραγματικό ολόκληρο μεγάλο πρόγραμμα. 7 δις ευρώ έφτασε το κόστος του ίτερ Οι επιτροπέ ερεύνησαν την αιτία του προβλήματο αυτού, αυτή της αύξησης του κόστους. Υπήρξε μια κοινή αντιπροσωπεία. που πήγε στον πυρηνικό αντιδραστήρα ο οποίος δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ΙΤΕΡ. Οι αιτίε έδειξαν σαφώς ότι όπω γίνεται συνήθω σε τέτοιε διαδικασίε, υπάρχει μια μελέτη που αξιολογεί το κόστος και μετά όταν ε, υπάρχει το εργοτάξιο το συγκεκριμένο, είναι συγκεκριμένα και τα, το κόστος μεταφοράς, μετά όσο εξελίσσεται το πρόγραμμα το κόστος γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο, ίσως προκύπτουν κόστη που δεν είχαν υπολογιστεί από πριν. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απαντηθεί είναι το ποιος ε, δημιουργεί αυτό το έξτρα κόστος. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, δυνατότητα ε, που μας, έδειχνε, που μας έδινε η, ε, ο τομέας της έρευνας στην Ένωση Είπαμε ότι το 2030 θα, ουσιαστικά θα πραγματονόταν αυτό το έργο γιατί τότε θα μπορούσε να λειτουργήσει και με βάση τεχνολογία. Γι' αυτό λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο το ερώτημα αυτό που και στο Κοινοβούλιο και στα κρατημέλη του Συμβούλιο για το πώ δηλαδή θα συνεχίσουμε να α, χρηματοδοτούμε το ίτερ γιατί έπρεπε να έχουμε σαφή καταγραφή του κόστους. Αυτό λοιπόν το διεκπαιρώσαμε αλλά παρόλα αυτά παραμένει το ερώτημα και αυτό ήταν το κίνητρο για μένα για να, κάνουμε για να γίνει αυτή η μελέτη. Καταρχάς, Έχουμε υπόψη μας όλους τους ε, κινδύνους. Δεύτερον, από πλευρά ε, οργανωτικής, πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Και η μελέτη ελπίζω ότι θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς ε, που λένε ότι οι κακές ειδήσει είναι τελικά καλές ειδήσει. Ε, όταν έχουμε καλές ειδήσει, ναι, αυτές είναι καλές ειδήσει. Οπότε ε, δεν θέλω βεβαίω να προκαταλάβω αυτά που θα πούνε οι συνάδελφοι από την Ernest Young, αλλά δείχνει αυτό ότι ε, πρέπει να ελέγξουμε το κόστος και από την τεχνική του πλευρά. τα πράγματα έχουν εξελιχθεί θετικά. βεβαίω πάντα υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. Υπάρχουν κάποιε συστάσει έτσι ώστε να υπάρξει υλικό και για τη δική μας συζήτηση με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Θα έχουμε υλικό λοιπόν για τροπολογίες, για την υποβολή του προπολογισμού, για την απαλλαγή για το ίτερ, για τις ε, σχετικές υπηρεσίες της Κομισιόν, οι οποίες εκπροσωπούνται. Χαίρομαι λοιπόν ε, για την επόμενη παρουσίαση που θα ακούσουμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή που προκάλεσε αυτή την ε, μελέτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. του δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι για την έρευνα. Ήθελα να τονίσω η Ernst και Young είναι μια, ένας φορέας που περιέχει μια ομάδα που ασχολείται με τις δημόσιες πολιτικές και έχει κάνει αυτές τις εργασίες. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάιερ για την υποστήριξή του. Η έρευνα γίνεται μεταξύ Ιουνίου 2012 και Φεβρουαρίου 2013 και ήταν μια ανάλυση της ε, άσκησης ε, ελέγχου του κόστους του F4E ε, που είναι μια κοινή προσπάθεια ανάπτυξης της ενέργειας από σύνδεξη και που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα ITER και επομένως ε, είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, δεν αναλύουμε το συνολικό κόστος του σχεδίου ITER στο σύνολό του. Είχαμε κάπου 42 συνεντεύξεις για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλους τους εμπλεκομένους στο F4E. Ε. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και το προσωπικό της F4E ε, που ήταν διαθέσιμο για αυτές τις επαφές, του εκπροσώπους κομισιών, των Κατών μελών και τους βουλευτές που ασχολήθηκαν για τα θέματα αυτά σε σχέση με τη συγκριτική ανάλυση benchmarking που μας επέτρεψε να δούμε και ποια είναι η κατάσταση σε αντίστοιχους φορείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για αυτήν την, ε, ε παρουσία, ε, και δίνω το λόγο τώρα στους ε, υπευθύνου. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ταχαίως, εντάχει, θα σας παρουσιάσω λιγάκι το γενικό πλαίσιο της μελέτης μας, παρά το γεγονός ότι τα βασικά στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί από τον κύριο Γκάιερ και από την συνάδελφόν μου. Το σχέδιο ITER είναι ένα σχέδιο επιστημονικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, το οποίο συνενώνει επτά εταίρους, επτά ε, χρηματοδότες για το σχέδιο αυτό και έχει σαν στόχο να καταδείξει το εφικτό της χρήσης της πυρηνικής σύνδεξης ως πηγής ενέργειας. Και αυτά απλώς μια επενθύμηση, οι επτά εταίροι που εμπλέκονται στο ΙΤΕΡ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία. Όπως είπε ο κύριος Γκάιερ, τα πρώτα χρόνια του σχεδίου αυτού η ΤΕΡ είδαμε μια πραγματική έκρηξη του κόστους για να επαναλάβω αυτά που είπε πράγματι οι αρχικές εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για το σχέδιο ΙΤΕΡ προέβλεπαν ένα συνολικό κόστος 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το σχέδιο και 2,7 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταχαίως διαπιστώσαμε ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό φρούδες αυτές οι εκτιμήσεις. Ξεπεράστηκαν οι αρχικές λοιπόν εκτιμήσεις μια δεύτερη εκτίμηση το 2008 έθεσε το κόστος σε, το συνολικό κόστος σε 7,2 δισεκατομμύρια και 7,2 δισεκατομμύρια μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 5,9 δηλαδή για την Ευρατόμ και 1,9 για τη Γαλλία. Μετά από πολύπλοκες διαδικασίες το 2010 υπήρξε μια συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να τονίσει και πάλι το ότι συμμετέχει και δεσμεύεται για την επιτυχία του εγχείρηματος αυτού και δέχτηκε να αυξήσει τη συμμετοχή της σε 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ με αυτό το 6,6 ως ανώτατο όριο <clears throat> για την επίτευξη της πρώτης φάσης του σχεδίου αυτού μέχρι το 2020. Εδώ στο γράφημα αυτό βλέπετε με ποιο τρόπο η υπηρεσία F4E, ε, Fusion for Energy δηλαδή, είναι ο φορέας ο ευρωπαϊκός για το σχέδιο ITER και είναι η διαδραστική επιφάνεια μεταξύ του ITER, του επιστημονικού τμήματος του σχεδίου αυτού και των βιομηχανικών φορέων ή των ερευνητικών εργαστηρίων που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Κατά ως εκ τούτου η F4E ε είναι αυτή η οποία διαχειρίζεται την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχέδιο αυτό. Βλέπετε εδώ κάποια αριθμητικά στοιχεία τα οποία τοποθετούν κάπως καλύτερα τη δράση της F4E, ε, F4E. Ε, ε, Το 2011 υπήρξε δέσμευση πιστώσεων ύψους 492 εκατομμύριων ευρώ και πιστώσεις πληρωμών 264 εκατομμυρίων ευρώ 99,7 του ποσού που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό δηλαδή πλήρης δέσμευση σχεδόν των ποσών αυτών Εάν τώρα ρίψουμε ένα βλέφαρο στο γράφημα που είναι δίπλα, βλέπουμε ένα πρώτο δίκτυ αποτελεσματικότητας του φορέα F4E, ε, γιατί βλέπουμε ότι τα χρόνια πριν από το 2011 το κόστος του λειτουργικού προϋπολογισμού έχει εκραγεί από 167 σε 611 εκατομμύρια ευρώ ενώ συνάμα το διοικητικό κόστος παραέμεινε ταπεινό σε λογικές αναλογίες, η αύξηση ήταν πολύ μικρότερη. <clears throat> Τα τέσσερα αυτά χρόνια είχαμε πραγματικά μια βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του φορέα που μπορούμε να καταμετρήσουμε με το γράφημα αυτό. Μετά από αυτήν την ταχεία παρουσίαση εισαγωγικού χαρακτήρα μπορώ να σας παρουσιάσω τα έξι κύρια συμπεράσματα τα οποία προέρχονται από τη μελέτη μας. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι και το οποίο είναι ότι η αύξηση του κόστους του ΙΤΕΡ προέκυψε κυρίως σε επίπεδο σχεδίου, του σχεδίου αυτού καθεαυτού και βασίστηκε σε παράγοντες οι οποίοι διέφευγαν της δυνατότητας ελέγχου της F4E. Ε. Όπως είπα και προηγουμένως, η F4E ε δεν είναι παρά μόνο ο φορέας ο οποίος διαχειρίζεται την εφαρμογή της ενωσιακής συνεισφοράς, αλλά τα τεχνικά στοιχεία διαχείρισης του προγράμματος προχώνται από τον φορέα ITER, και όλες οι προμήθειες υλικού και υπηρεσιών έρχονται από το ΙΤΕΡ, η F4E ε μεταβιβάζει αυτές τις ε, διαδικασίες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που απαιτεί το ΙΤΕΡ. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι η F4E ε ειναι μια ιδιότυπος sui generis οργάνωση μέσα στο στερέωμα των ευρωπαϊκών φορέων και λειτουργεί σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο. Και έχει πολύ μικρό έλεγχο σε αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον και έχει πολύ μικρές δυνατότητες να περιορίσει την αύξηση του κόστους και να εξασφαλίσει μια βελτίωση της σχέσης κόστους-οφέλους διότι δεν έχει τον απαραίτητο έλεγχο στο περιβάλλον της. Τρίτον, η F4E ε αντιμετώπισε και πρώιμες δυσκολίες, οι οποίες προέκυψαν πολύ ενωρίς και αφορούσαν ιδιαίτερα τις διαχειριστικές δομές και την διακυβέρνηση του φορέα αυτού και το συμπεράσμα μας στο θέμα αυτό είναι ότι αυτά τα προπατορικά προβλήματα έχουν τώρα διαπιστωθεί και εντοπιστεί, έχουν αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό και βέβαια είναι νωρίς για να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα σε σχέση με τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση του φορέα αυτού, αλλά φαίνεται σαφώς ότι το έδαφος έχει ενισχυθεί για τον φορέα αυτό και πιστεύουμε σήμερα ότι η F4E ε έχει αρκετά στερεές δομές για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις και τις αποστολές του μέλλοντος. Τέταρτο συμπέρασμα. Υπάρχει δυνατότης βελτίωσης. Υπάρχουν τομείς στους οποίους έχουμε εντοπίσει δυνατότητες βελτίωσης, αλλά πρέπει να πω ότι η δυνατότητα διαχείρισης του κόστους και περιορισμού του κόστους από το φορέα μας είναι οριακού χαρακτήρα. Αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιους τομείς όπως οι διαδικασίες δημοσίων αγορών, η πολιτική ανθρωπίνου δυναμικού, και ο εσωτερικός έλεγχος και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του φορέα μπορεί να υπάρξει κάποιο, κάποια βελτίωση. Πέμπτο σημείο. Πρόκειται για το πρόβλημα της ικανότητας του φορέα αυτού να αντιμετωπίσει τα αστάθμητα και απρόβλεπτα γεγονότα. Όπως είπα προηγουμένως, μας φαίνεται στον τομέα αυτό ότι η απλή μορφή διαχείρισης του κόστους από το φορέα μας δεν θα του επιτρέψει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των αστάθμιτων γεγονότων μόνο με τον περιορισμό του κόστους είναι επομένως σε μια κατάσταση επισφαλή και είναι ευάλωτε στην πολιτική αβεβαιότητα η οποία μπορεί να θέσει να αφιβόλω το σχέδιο αυτό και επίσης από την χρηματο τη δημοσιονομική μάλλον αβεβαιότητα που περιστοιχίζει αυτό το σχέδιο. Το τελευταίο συμπέρασμα της μελέτης μας έχει να κάνει με την δυνατότητα συγκριτικών μελετών, benchmarking, που είναι ένα από τα θέματα της προβληματικής της μελέτης μας και για μια ακόμα φορά ο μοναδικός χαρακτήρας του φορέα F4E μας οδηγεί ακόμα στο συμπέρασμα ότι μια διαδικασία benchmarking δεν θα ήταν εύστοχη λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν συγκρίσιμες δομές από την, με την F4E και το να υπησέλθουμε σε αυτή την πρόσθετη άσκηση benchmarking ενώ ο φορέας αυτός έχει περάσει διάφορες μορφές ελεκτικού χαρακτήρα, λογιστικό έλεγχο κτλ. και τα λοιπά και παρακολούθηση θα ήταν μια ε, χωρίς ε, περιεχόμενο άσκηση που δεν θα ωφελούσε σε τίποτα. Έχουν παρουσιάσει αυτά τα γενικά συμπεράσματα, θα, θα θελήσω τώρα να δώσω το λόγο στον συναδελφό μου, ώστε να αναπτύξει περαιτέρω τα απορίσματα και τις συγκεκριμένες συστάσεις που εξέρχονται από την μελέτη μας. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα αγγλικά τώρα. Το συμπέρασμα 4, όπου εντοπίσαμε διαφορετικούς τομείς, όπου μπορούσε να επιτελεστεί πρόοδος, παρά τους περιορισμούς και τις πιέσεις. Οι συνάδελφοι ήδη τα έθιξαν. Ο πρώτος τομέας, ο τομέας που ήταν ο πλέον εμφανής και ο μόνος που πραγματικά έχει την ικανότητα να επιτρέψει την αντιμετώπιση πηγόντων και το χτίσμα μιας τέτοιας ικανότητας είναι οι δημόσιες προμήθειες. εδώ είναι περιορισμένο και επικίνδυνο πεδίο, αλλά υπάρχουν τρία σημεία για τον έλεγχο του κόστους. Το πρόγραμμα F4E έχει δώσει δυνατότητα για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και συμμετοχή φορέων με μελέτες, εκπόνηση μελετών που μπορεί να επιτρέψει να καταλάβουμε καλύτερα την αγορά και να αντιμετωπίσουμε κινδύνους. Οι απειλές μπορούν να αναταχαιριστούν αποτελεσματικότερα. Το πρόγραμμα Fusion for Energy έχει πολύ αποτελεσματικά κινηθεί προ το βιομηχανικό κλάδο και ο βιομηχανικό κλάδο ο βιομηχανικός κλάδος ίδιος είχε προσαρμοστεί στις ανάγκες του προγράμματος και σα απαιτεί για τις δημόσιες προμήθειες. Αρκετά εγκαίρως ε, παρουσιάστηκαν, αρκετά γρήγορα μάλλον παρουσιάστηκαν ε, στην υλοποίηση του προγράμματο αδυναμίες. Κυρίως ως προς τον ε, προς τη διοργάνωση. Μπόρεσε όμως το Διοικητικό Συμβούλιο, ακριβώς επειδή παρουσιάστηκαν γρήγορα οι αδυναμίες, να πάρει στρατηγικές αποφάσεις και να τις αντιμετωπίσει. Βέβαια, παρά την καλή διαχείριση του προγράμματος που παρατηρήσαμε, χάρη στις ενέργειες των συμμετεχόντων, οι διαδικασίες ήταν κάπως πρόχειρες Χρειάζεται ένα πρόγραμμα εργασίας ετήσιο με ρητές εξηγήσεις και λεπτομέρειες για το τι θα γίνει τα ερχόμενα χρόνια. Κάτι που να αναφέρει τις αναγκαίες αλλαγές και ένα περιθώριο εξαμήνου. Η μελέτη Ernst Young, ένα από τις πρώτες άνοιξε το δρόμο για τη δική μας μελέτη και επικεντρώθηκε στην ανάγκη να βελτιωθούν οι ορισμοί περιορισμού στατικών μάλλον περιορισμού του κόστους οι αξιολογήσει των στατικών αυτών και με, ενδεχόμενους, με τη χρήση ενδεχόμενων ποσοτικών δικτών. σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη και τη συμφορά τους στο F4E, αυτό τέθηκε ως ερώτημα στην αξιολόγηση αυτή καθεαυτή και θεωρήσαμε ότι τα πρωτόκολλα δεν αρκούν, αυτά που ισχύουν για τα κράτη-μέλη, ώστε να έχουν άμεση συνεισφορά, μεγαλύτερη άμεση συνεισφορά στο πρόγραμμα. Μπορεί μάλιστα να προκύπτουν προβλήματα λόγω της δυσμενούς και προσωρινής θέσης στην οποία βρέθηκε το ε, F4E με την έλλειψη εργαλείου αντιμετώπισης επιγόντων. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι των κρατών μελών με τους οποίους συζητήσαμε κατέδειξαν τα εργαστήρια σύνδεξης των κρατών μελών ως μια δυνατότητα για την ε, τόνωση της συμμετοχής των κρατών μελών. Ιδίω από τη στιγμή που άρχισε να λειτουργεί το πρόγραμμα ITER, τα εθνικά εργαστήρια σύνδεξη γνώρισαν μείωση στον προπολογισμό του. Υπήρξαν υποσχέσει από τι εθνικέ αρχέ ότι αυτό θα αντισταθμιδιόταν μέσω δωρεών του F4A, αλλά αυτό δεν υλοποιήθηκε. Αυτή η διασύνδεση με τα εθνικά εργαστήρια σύνδεξη θα έδινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δυναμικό να υποφεληθεί από το Programmator. Αλλά είμαστε επιφυλακτικοί ως προς την αποτελεσματικότητα, τη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας ε, με την συμμετοχή των εργαστηρίων σύνδεξης. Υπάρχουν πολλοί νομικοί πραγματικοί δυσκολίες μεταξύ των οποίων ανταγωνισμός, κανονισμοί, το γεγονός ότι πολλά εργαστήρια δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κονδύλια για να φτάσουν στα ύψη των προσδοκιών του ΙΤΕΡ. Η υλοποίηση στην παρακολούθηση και το σύστημα ελέγχου. Ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια ιδίως από το 2011, με την αλλαγή της δίκησης. Το F4A, 4E, έδωσε στο βιομηχανικό αυτό κλάδο ε, συγκεκριμένα βασικά συστήματα μέσω εσωτερικής υποβολής εκθέσεων, συνεντεύξεων, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των δεδομένων. Βεβαίω, το έλεγαν ανέκαθεν οι συμμετέχοντες, το επόμενο στάδιο στο F4E θα ήταν η καλύτερη συμπερίληψη στοιχείων και άλλων προγραμμάτων. Το Fusion for Europe και ο συνδυασμός με τις δράσεις ITER οδηγούσαν σε παραλληλισμό δραστηριοτήτων. Χάρη σε δεμερείς συμφωνίες μεταξύ των επιχειρημάτων ε, ήταν το γεγονό ότι η συχνότητα των παράλληλων δραστηριοτήτων θα πρέπει να επανεξεταστεί προκειμένου να μην προβλήψουν περαιτέρω δημοσιονομικές πιέσεις. Τέλος, οι κανονισμοί προσωπικού ίσως να μην είναι εύστοχοι για το εφορί ο μακροπρόθεσμος δρόμος αποτελεσματικότητας που έχει στοχεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να μην συνάδει πλήρως με τις ανάγκες του προγράμματος σύνδεξη για την Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα καθημερινού χαρακτήρα, όπως το κόστος ζωής στη Βαρκελόνη. Δύσκολα μπορεί κανείς να προσελκύσει μέλη για τη διοίκηση με τα όσα ισχύουν εκεί. Αυτά είχα να πω για, τις συγκεκριμένες, για τα συγκεκριμένα ευρήματα της μελέτης. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Συζητήσαμε για το ΙΤΑΡ ήδη διαπιστώνω ότι είναι πολύ ευρέα τα, τα, τα αποτελέσματά σας. Ε, προφανώς ε, ε, ο συνδυασμός των ε, ενεργειών δεν λύνει πάντα το πρόβλημα. Το θέμα είναι που υπάρχουν κονδύλια για να εισρέψουν σε τέτοια προγράμματα και αυτό νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουν και η πυρηνική φυσική αλλά και άλλοι επιστήμονες τους πέφτει περισσότερος λόγος από εμάς τους ελεγκτές, τους οικονομολόγους. Βαλτσίτης, μετά ο Γκάιερ και ο Γιάνν Μιούλντερ έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω μαζί σας σε σχέση με το εύρος επιρροής του ίτερ. Βεβαίως, το πεδίο εφαρμογή θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και θα πρέπει να μιλήσουμε κυρίως για τη χρήση των κονδυλίων. Ο εισηγητής ανέφερε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να μας δείξει ότι πρέπει να λυθούν τα προβλήματα, αλλά αυτό που λέει ότι υπάρχει όλο και λιγότερη πολιτική βούληση για να χρησιμοποιηθούν ε, τέτοια προγράμματα. Αυτό προφανώς δημιουργεί κάποια ανησυχία. Και πριν από λίγο καιρό επισκέφθηκα μια μεγάλη ε, επιχείρηση η οποία επίσης ασχολείται με μεγάλα προγράμματα τα οποία είναι, ε, έχουν ε, κάποιες φάσεις και σε κάθε φάση του προγράμματος γίνεται και μια αξιολόγηση. Αυτή η, αυτή η επιχείρηση ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της γενετικής και είναι εξίσου περίπλοκη η δουλειά της όπως και η πυρηνική σύνδεξη. Λοιπόν, Ίσως ε, να βγαίνει το συμπέρασμα από εδώ ότι οι ε, στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτό μπορεί να ε, θέσει ένα αμφιβόλο και τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Βεβαίως εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων σε αυτό το θέμα, αλλά όλοι μας είμαστε κατά κάποιο τρόπο εμπειρογνώμονες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων. Γι' αυτό θα πρέπει αυτές ακριβώς τις ε, φάσεις των διαφόρων προγραμμάτων να τις εξερολογήσουμε και να δούμε τι γίνεται με τη στοχοθέτηση ε, για τα επόμενα χρόνια, από το 2013 στο 2015 ας πούμε. Ίσως θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε την εφαρμογή των διαφόρων φάσεων των προγραμμάτων. Μιλούμε για ε, πολιτική βούληση από τις ε, χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτή δεν υπάρχει, τότε το ελεκτικό συνέδριο ίσως να πρέπει να υποβάλει κάποιες ε, συστάσεις για την αξιολόγηση τέτοιων προγραμμάτων. <clears throat> Ευχαριστώ. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους ε, συναδέλφους από την Ένωση και και χαίρομαι που ε, συζητούμε το θέμα αυτό. Βεβαίως, η συγκρισιμότητα καθιστά ε, δύσκολο της, καθιστά δύσκολη την κατάσταση στην αγορά. Αυτές οι συσκευές δεν υπάρχουν, δεν έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και απ' την άλλη Νομίζω ότι για την Κομισιόν το ίτερ είναι έτσι σαν, σαν ένα σαν ο πίθος των Δαναών. Η ευθύνη για την διαχείριση των κονδυλίων παραμένει βεβαίως στο F4E και βεβαίως η πολιτική διαχείριση. Ίσως να μην ταιριάζει στις απαιτήσει που έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εγώ μέσω της ε, έρευνα είδα ότι αυτές οι συγκεκριμένε, πολύ συγκεκριμένε απαιτήσει που έχει το πρόγραμμα αυτό για, σε ό,τι αφορά την ε, ε, επιστημονική ή βιομηχανική εμπειρία των, του προσωπικού είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυαστεί με έναν ιστορικό κανονισμό ή με ένα οργανόγραμμα. Βεβαίω αυτό σημαίνει ότι κάπου θα πρέπει να γίνει κάποιο συμβιβασμό. Ή θα αλλάξει το οργανόγραμμα, που βεβαίω είναι θέσπατο και δεν αλλάζει, ή κάτι πρέπει να γίνει με το προσωπικό. Αλλά και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες στην ε, ε, ε, ποιότητα της εκτέλεσης του προγράμματος. Και το θέμα των παράλληλων δραστηριοτήτων. Και αυτό είναι ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Θα μπορούσαμε βεβαίω να ακούσουμε την Κομισιόν από αυτού, αλλά αν μέσω Twitter που είναι η ομπρέλα, μπορεί το Fusion for Europe να αναλάβει κάποιες παράλληλες δραστηριότητε, τότε εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι υπάρχουν κάποιες συμβάσεις που μπορεί να έχουν σχέση με την ε, σύνδεξή αλλά δεν συνδυάζονται προς το παρόν με την εκτέλεση των προγραμμάτων. Και αυτό επηρεάζει το κόστος. Αν λοιπόν κάποιος ενδιαφέρεται να αναλάβει αυτές τις ε, δραστηριότητες, ίσως εμείς ως ε, αρχή προπολογισμού να θέσουμε το ερώτημα ποιος θα καταβάλει το κόστος όλων αυτών. Επίσης από τη μελέτη είδα που πρέπει να παρέμβουμε σε πολιτικό επίπεδο. Βεβαίω αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το, κάνουμε με, πρέπει να το συζητήσουμε με ε, τις διάφορες υπηρεσίες. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μούλδαλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τα 30 χρόνια ακούμε ότι η σύνδεξη θα γίνει πραγματικότητα κάθε φορά που μας το λένε για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό το λέμε κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια. Και αρχίζει να φαίνεται δύσκολο αυτό. Ελέγχθη ότι ο φορέας σας δεν μπορεί να προβλέψει το κόστος και οποιαδήποτε μείωση κόστους θα είναι περιορισμένη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Έχουμε ένα προϋπολογισμό για το ΙΤΕΡ για τα επόμενα 7 χρόνια. Αλλά μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις κόστους για οποιοδήποτε λόγο. Είναι δυνατόν να δώσετε κάποια πρόβλεψη για το αν είναι ρεαλιστική πιθανότητα η πυρηνική σύνδεξη να γίνει κάποτε μία πηγή ενέργειας και είσαστε πεπισμένος ότι οι προβλέψει που έχουμε στον προϋπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια θα είναι ο πραγματικός προϋπολογισμός που θα απαιτηθεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Ακολουθεί η κυρία Μόνικα Χόλμαερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ιδιαίτερος πολύπλοκο ερευνητικό πρόγραμμα. Είναι πολύ φιλόδοξο, αλλά όπως είπε και ο κύριος ε, Γκάιγερ, είναι ένα απόλυτα μοναδικό σε σχέση με τη μορφή του πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν συγκρίσιμα τέτοια εγχειρήματα γιατί αυτό καλύπτει πάρα πολλούς κλάδους της επιστήμης. Εγώ έχω αντιμετωπίσει και τα θέματα Twitter και του Fusion for Energy. Το πρόβλημα βέβαια δημιουργείται και από το γεγονός ότι πρέπει να συνεργαστούμε με ένα διεθνές consortium και είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και επίσης και η οργάνωση της κατανομής των αρμοδιοτήτων και όλα αυτά δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σαφή. Όταν έχουμε τόσες πολλές χώρες και τόσες πολλές υπήρους δεν είναι εύκολο το εγχείρημα αυτό και ο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων δεν είναι ιδιαίτερα εύκολος για να μπορέσει να υπάρξει μια άκοπη συνεργασία για όλα αυτά τα θέματα. Όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχω την εντύπωση ότι στο Fusion for Energy Γίνονται πολλές προσπάθειες για τις ε, δικές της αρμοδιότητες της F4E ε. και σε μεγάλο βαθμό μπορεί αυτός ο φορέας να αντιμετωπίσει τις ε, διαδικασίες δημοσίων αγορών. Βέβαια αυτό γίνεται σε μήκος χρόνου. Είναι μια μακροχρόνια και μακρόπνοια διαδικασία αλλά μόνο τώρα έρχεται το πρόγραμμα ITER και το f 4 σε ένα στάδιο που γίνεται ενδιαφέρον, που χτίζονται εγκαταστάσεις, όπου γίνονται οι πρώτες ε, λειτουργίες προγραμμάτων σε πραγματικό ερευνητικό επίπεδο. Είναι τώρα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε την πιο μεγάλη πρόκληση για να υποστηρίξουμε τα σχέδια αυτά. Αυτό το οποίο για μένα είναι σημαντικό είναι να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία, η οποία δίνει τα περισσότερα χρήματα σε αυτήν την ε, οργάνωση και δεν είναι προβλήματα ενδογενή στο Fusion Forensics, στο F4E, αλλά προβλήματα στο ITER τα οποία προκαλούν δυσκολίες μέσα στο F4E. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να διεκδικήσει μια πιο ισχυρή θέση μέσα στο ΙΤΕΡ, γιατί δεν αρκεί το γεγονός ότι από τη μια μεριά η Κομισιόν έχει μονάχα μία έδρα στο Συμβούλιο του ΙΤΕΡ, από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να εξασφαλίζει την χρηματοδότηση του f 4 ε Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες δυνατότητε επιρροής μέσα στο ΙΤΕΡ ως ε, σύνολο. Δεύτερον, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να προσπαθήσει το F4E ε να βελτιώσει τις δομές για τις ε, δημόσιες αγορές και να τις προσαρμόσει στις νέες βιομηχανικές ε, συνθήκες. Υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι υπήρξαν σε πολλές περιπτώσεις προβλήματα αστικής ευθύνης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη πιο προσεκτικά στις διαδικασίες δημοσίων αγορών, διότι μιλάμε για αγορές οι οποίες είναι πραγματικά εξειδικευμένου χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν όλα αυτά τα στοιχεία πριν από την ε, προκήρυξη των διαγωνισμών και όχι αφού έχει γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού και χρειάζεται να γίνουν αλλαγές. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει από το F4E ε θα πρέπει να μεταφερθούν και στο ε, συνολικό πρόγραμμα ITER. Γιατί το ITER είναι ένα σχέδιο στο οποίο δεν έχει καμία δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγξει το τι γίνεται και το κόστος. Νομίζω ότι αυτός δεν είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Η Κομισιόν μας έχει εξηγήσει ότι φυσικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι κάτω από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας και δεν θα είναι τελείως ανεξέλεγκτα ε, και να αποφασίζονται από το ίτερ. Αλλά βλέπουμε ήδη τις δυσκολίες για το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο διεθνές κονσόρτσιουμ το οποίο δεν δεσμεύεται από τους κανόνες και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχει την δικιά του ίδια δυναμική. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει <clears throat> να εξασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα που δίνουμε θα πρέπει να έχουν και ένα αντίκρισμα στο ρόλο μας μέσα στον φορέα του ΙΤΕΡ τον ίδιο. Ναι, κατανοώ. Επειδή τελειώνει ο χρόνος, θα ήθελα να ζητήσω στον κύριο, από τον κύριο Ρούμπικ να κάνει μια τελευταία παρέμβαση πρώτου δώσουμε το λόγο και στην Κομισιόν και στους ε, εκπροσώπους της Ernest αλλά και Young. Το ερώτημα είναι πώς θα προχωρούσε αυτό το πρόγραμμα αν δεν υπήρχε καμία υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ήταν μονάχα η διεθνή σε αυτή η εταίρη. Ωραία. Δίνω τώρα το λόγο στην Κομισιόν, παρακαλώ. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. I was hoping uh, as Ήλπιζα ως ε, διευθυντής να μιλήσω εγώ πρώτος. Μπορώ, ευχαριστώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Ernest Young για την πολύ καλή έκθεση που έκανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ λίγες ε, δυνατότητες. Μπήκατε σε βάθος σε ένα πολύ περίπλοκο θέμα και θέλω επίσης να καταγραφεί ότι εδώ ε, ασχολούμαστε με κάτι που είναι πολύ τεχνικά δύσκολο και οργανωτικά επίσης πολύ δύσκολο. Και για να σας εξηγήσω γιατί ακριβώς το κυνηγάμε αυτό, πρέπει να σας πω ότι αυτή η τεχνολογία δεν είναι μια οποιαδήποτε τεχνολογία. Η ενέργεια είναι στην καρδιά της οικονομικής ευημερίας των χωρών μας. Υπάρχουν λίγες, λίγα είδη ενέργειες που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να κάνουμε τις μεγάλες περικοπές, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που θέλουμε να κάνουμε στα επόμενα 50 χρόνια. Το Fusion for Energy είναι πραγματικά εξαιρετικό σε αυτό το τομέα. Μόλις ε, καταφέρουμε να κάνουμε τη σύνταξη, θα, τη θα έχουμε κάτι που μπορεί να βοηθήσει τις βιομηχανοποιημένες χώρες σε τεράστιο βαθμό και επίσης δεν είναι μια προσωρινή πηγή ενέργειας, είναι μια πηγή που θα κρατήσει μέχρι να καταστραφεί ο κόσμος. Είναι λοιπόν συγκλονιστική αυτή η εξέλιξη. Οι, όλες οι χώρες ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τη βιομηχανική λοιπόν, δυνατότητα, τις τεχνικές αποδομές ως προς αυτό. Η Ευρώπη είναι ε, η πρωτοπόρα σε αυτό το τομέα. Η Κίνα, η Ιαπωνία θα ήθελαν να μας προλάβουν και να βγουν πρώτες. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε και να επιτύχουμε αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα δημιουργήσει τις εγκαταστάσεις για να γεμίσει το κενό που υπάρχει μακροπρόθεσμα όταν το Fusion for, Industry γίνει, ε, Fusion for Energy γίνει πραγματικότητα θα τα πράγματα θα είναι σαφω καλύτερα. Αλλά προ το παρόν είναι τεχνολογία έχμη, αυτή, είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και έτσι οδηγούμαστε σε, ένα πολύ, σε μια πολύ περίεργη δομή όπου υπάρχουν διάφορα διασυνδεόμενα στοιχεία τα οποία ε, εξελίσσονται και στην Ευρώπη αλλά και στους εταίρους της. Βεβαίως ως βιομηχανία δεν θα βρώσε κανείς έτσι αλλά λόγω ακριβώς και των, ε, των ε, δυνατοτήτων που έχει η, η τεχνολογία προχωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, έχει λοιπόν πρέπει να τις ε, προωθήσουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε και την ε, βιομηχανία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ε, μεγάλη διασύνδεση και με την Ίτερ, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί 7 υπηρεσίες οι οποίες δεν παρέχουν απλώς αλλά σχεδιάζει η Ευρώπη και το πώς θα λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες. Υπάρχουν λοιπόν πολύ περίπλοκες διασυνδέσεις και κατά συνέπεια βλέπουμε ότι οι απαιτήσει αυξάνονται συνεχώς. Για παράδειγμα, όταν έγινε το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, οι απαιτήσει προφανώς αυξήθηκαν. Αυτό οδήγησε σε επιπλέον απαιτήσει που προφανώς αυξάνουν το κόστος. Παρά αυτέ τις αυξημένε απαιτήσει. εξακολουθούμε να διατηρούμε μόνο κάποιες από τις δυνατότητες που είχαμε. Βεβαίως θέλουμε να ε, ε, μειώσουμε το κόστος όσο γίνεται περισσότερο. Το διαπίστωσε και η Ανεστιγιάννη και αυτό και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει αυτό το διάλογο με τη βιομηχανία ενεργά έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά στα βιομηχανικά πρότυπα. Και βεβαίως έτσι ε, παρακλίνουμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε στην αρχή να ακολουθήσουμε την Κομισιόν. Οπότε τώρα ακολουθούμε το δρόμο της βιομηχανίας. Αυτό ίσως σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση σε σχέση με τους κανόνες βάσει των οποίων λειτουργούμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι στις 6.30 πρέπει να σταματήσουμε. Είναι 6.30. Λυπούμε γι' αυτό λοιπόν. Ένα λεπτάκι θα σας δώσω. Fusion Laboratories is key. Τα εργαστήρια σύνδεξης επίσης είναι σημαντικός παίκτης γιατί εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γνώση σε ό,τι mm. αφορά το, Europe, το Fusion for Europe. Υπάρχει διασύνθεση βεβαίως με αυτά και θεωρούμε ότι θα υπάρξει τεράστια σχέση και με την ε, προμήθεια σε ό,τι αφορά το, ότι θα είναι, ε, τα εργαστήρια θα είναι οι εταίροι που θα ασχολούνται ακριβώς ε, άμεσα με το θέμα αυτό και θα μπορέσουμε έτσι να διευκολύνουμε την ε, μεταφορά γνώση από τον ε, δημόσιο τομέα στη βιομηχανία. Έχω πάρα πολλά να πω ακόμα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Και τώρα, επειδή ήταν πολλές ερωτήσεις, όσο κρατώ πιο γρήγορα, πολύ σύντομα να δώσω κάποια στοιχεία για όσα εφήγησαν ιδίω από τον κύριο Μούλτερ. Απλώς να θυμίσω ότι η μελέτη μας αφορούσε τον έλεγχο του κόστους της Fusion for Europe. Στα συμπεράσματά μας είπαμε ότι το κόστος που προκύπτει, προκύπτει από το σχέδιο, από το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. Ο οργανισμός, το πρόγραμμα δεν έχει έλεγχο για το κόστος αυτό. Όσο αφορά την επιστημονικό ή την τεχνική διάσταση, τη δημοσιονομική προσαρμογή που προκύπτει από το κόστος, η μελέτη μας δεν το κάλυψε αυτό και δεν μπορούμε να σας δώσουμε επιπλέον στοιχεία. Για τα υπόλοιπα σημεία που έθιξαν ε, οι υπόλοιποι βουλευτές, κυρίως ο κύριος Μούλτερ, η προσαρμογή των διαδικασιών των δημοσίων προμηθειών είναι κάτι που περιλαμβάνεται στις συστάσεις της έκθεσης. Θα χρειαστεί καλύτερη μόχλευση για τον έλεγχο του κόστους λειτουργίας του οργανισμού. Ήσασταν πάρα πολύ συμπαγείς και σύντομος. Προφανώς θα πρέπει να συζητήσουμε τη συζήτηση σε άλλους χώρους. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε. Ο εισηγητής δεν ζητά το λόγο περαιτέρω. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους, ιδιαίτερα την Earth και Young για την παρουσίαση αυτής της μελέτης, αλλά και την F4E και την Κομισιόν. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επανέλθει στα θέματα των εμπειρογνωμόνων, αυτά και να συζητήσει περαιτέρω το θέμα αυτό. Κλείνει λοιπόν η συνεδρίαση της Επιτροπής ελέγχου του προπολογισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τους, και τη γραμματεία και το, τους εκπροσώπους του Ελεκτικού Συνέδριου και τις κοπέλες που μεταφράζουν.